E Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Θα διαβιβάζω ότι έλαβα από τις αρμόδιες ρουμανικές αρχές έτοιμα ανάκλησης της ασυλίας ε, του συναδέλφου Αντριάν Σεβερίν αίτημα το οποίο απεστάλλει από την Γενική Διεύθυνση κατά της Διαφθοράς της Ρουμανίας βάσει του άρθρου 6 παραγράφου 2 του κανονισμού μας. Το αίτημα ανάκλησης της ασυλίας ε, παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή που είναι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Έλαβα επίσης αίτημα... Παρακαλώ κύριε Αλφάνο. Κύριε Αλφανό, ε, κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία, θα ήθελα να μου δώσετε λίγα λεπτά για να υπενθυμίσω στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πριν από δύο χρόνια είχαμε το σεισμό στην Άκουιλα όπου ε, χάθηκαν 280 ζωή και τραυματίστηκαν πάνω από 1.200 άτομα. Θα ήθελα ε, γι' αυτό το λόγο να αποστείλω σήμερα σε όλους τους ευρωβουλευτές ένα βίντεο το οποίο γυρίστηκε στις 6 ε, Ιανουαρίου στην Άκουιλα. Καλώ όλους τους συναδέλφους να το δουν διότι οι πολίτες της Άκουιλα περιμένουν ακόμα την στεναρή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Αλφάνο. Το είχα υπενθυμίσει και εγώ στην πρωινή συζήτηση ε, το τραγικό αυτό γεγονός. Ε, καλώς ε, κάνατε και το υπενθυμίσετε ενώπιον όλων των Ευρωβουλευτών. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Σασόλη. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Εχθές το βράδυ είχαμε μία ακόμα τραγωδία στη Μεσόγειο, μετανάστες οι οποίοι είχαν φύγει από τη Βόρεια Αφρική χάθηκαν ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ιταλία και την Ευρώπη. Έχουμε 130 αγνοούμενους, έχουν ε, ήδη 20 πτώματα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για άνδρες, γυναίκες, παιδιά και όχι μόνο για αριθμητικά στοιχεία. Φτάνει πια με τις ε, δισταγμούς, ε, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη πρέπει να δράσουν. Η Ευρωπή της Δημοκρατίας θα πρέπει να εκφράσει τη λύπη της για το θέμα αυτό και θα ήθελα να ζητήσουμε από την Ολομέλεια να τηρήσει ενός λεπτού σιγή προς τιμήν των θυμάτων της μετανάστευσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σασόλη. Βεβαίως και θα ικανοποιήσω το έτοιμά σας. Πριν να ζητήσω όμως να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για να υπενθυμίσουμε τα θύματα αυτά, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ταβάρες που ζήτησε να μιλήσει για το ίδιο θέμα. Thank you, President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ενημερωθήκαμε ότι ένα, μια, ε, ένα πλοιάριο από την Λιβύη ε, πνίγηκε και από όσων ξέρουμε χάθηκαν 150 ζωές. Σύμφωνα με την συναπόφωση, εμείς ε, στις αρχές του χρόνου έχουμε προβλέψει μηχανισμό έκτακτο για να μπορέσουμε να δεχόμεθα τους ε, μετανάστες αυτούς, αν υπήρχε πόλεμος όπως η Σιβία. Αυτό το θέμα ε, της συναπόφασης είναι ένα θέμα που τρενέδε και ένα χρόνο. Τον προηγούμενο μήνα με προφορική ερώτηση είπαμε πρόκειται για ανθρώπινες ζωές στο Συμβούλιο. Είναι σημαντικό. Και σήμερα αναμφισβήτητα το διαπιστώνουμε αυτό το πράγμα. Καλώς, ευχαριστώ. Κατόπιν αιτήσεως του συναδέλφου σας όλοι και νομίζω ότι ούτως ή άλλως μιλούσε εξ ονόματος όλων να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για να υπενθυμίσουμε ε, το χαμό των ε, απόψινων θυμών. Prego. Prego, Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Πρέγω. Ευχαριστώ. 20 δευτερόλεπτα απλώς και μόνο κύριε Πρόεδρε για να ακουστεί μία φωνή όχι πολιτικά ορθή. Εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι εξαιτία των απατηλών ελπίδων που δίνεται στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή λέτε ότι είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχθούμε όλους εδώ πέρα. Είστε λοιπόν αποκλειστικά υπεύθυνοι. Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Γιατί Έκθεση Γεντρεζεύσκα. Παρακαλώ, ησυχία, να ψηφίσουμε. Κυρία Μουσκαρδίνη, παρακαλώ. Παρακαλώ, σύντομα κυρία Μουσκαρδίνη. Ζητούσα το λόγο εδώ και κάμποση ώρα, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσα λεπτά συγγύης θα πρέπει να τηρήσουμε ακόμα προτού καταλήξουμε σε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση. Δεν είναι ώρα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση η οποία έγινε και χθες για το ίδιο ζήτημα. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Βάσει της απλουστευμένης διαδικασίας με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία.